η επιδότηση αυτή θα πρέπει να είναι ισότιμη για όλους. Τελειώνω, μπορείτε να αναπνεύσετε. Τάσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι άριστη, δεν είναι τέλεια, ούτε και θα είναι στο μέλλον. Αλλά είναι το καλύτερο πόσα θα μπορούσα να φανταστώ. Στην Ευρώπη για εκατοντάδες, χιλιάδες θα έλεγα χρόνια, η διαφορές ρυθμιζόντουσαν ε, με την δύναμη του πιο ισχυρού. Ποιος είναι ο πιο ισχυρός, αυτός επικρατεί, ο πιο αδύναμος, α, κρίμας, πρόσεχε. Τώρα πια εργαζόμαστε με διαφορετικό τρόπο, με έναν τρόπο που είναι καλύτερο από οποιονδήποτε άλλο είχαμε φανταστεί ποτέ στην ιστορία μας. Αυτή τη στιγμή συνεργαζόμαστε και αποφασίζουμε ε, με δική μας βούληση και με την επιθυμία των πολιτών μα. Κάποιο μπορεί να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά το Brexit αποδεικνύει πόσο δύσκολο είναι αυτό. Παρ' όλα αυτά, αποτελεί μαρτυρία του πώ λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η καλή θέληση και η, η συνένεση να παραμείνουμε σε μια Ευρώπη των 27 αποτελεί μαρτυρία και απόδειξη ότι είμαστε πεπισμένοι πως μέσω συζήτησης, μέσω του διαλόγου μπορούμε να παραμείνουμε ενωμένοι και να προχωρήσουμε χωρίς ε, να χρησιμοποιούμε βία, χωρίς να προσφεύγουμε στη βία. Μιλώντας ο με τον άλλο. Τώρα για το μέλλον. Συνοψίζοντας θα έλεγα ότι πρέπει να ενισχύσουμε τα βασικά. Την ενιαία αγορά, να καταργήσουμε τα, τους να ελέγξουμε καλύτερα τα εξωτερικά μας σύνορα, να μειώσουμε τον, την απειλή της ανεξέλεγκτης ε, μετανάστευσης, ε, ευφύης μετάβαση στι ε, ε μορφές ενέργειας, ε, ενίσχυση της ασφαλείας μας, όχι μόνο στο στρατιωτικό σκέλος, αλλά και στην ασφάλεια της πληροφορίας. Μην πολεμάτε τους λαϊκιστές. Αντιμετωπίστε την ουσία και τον λόγο της αιτία της ανησυχίας των πολιτών. Θυμηθείτε το μύθο αυτό του Εσώπου ε, με τις βέργες που είναι δύσκολο να τις πάσει κανείς όταν είναι μια θυμονιά. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να είναι ισχυρός παίκτη στην, ε, στον κόσμο και έχουμε βασικές αξίες ελευθερία, δημοκρατία, κράτος δικαίου και αυτές θα πρέπει να προβάλλουμε και στις άλλες χώρες του κόσμου. Ευχαριστώ. Ε, είστε πολύ δημοφιλής, ε, αγαπητέ κύριε Κριστιανής. Αγαπητέ Κριστιανής. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Ζαν Κλοντιούν, και έχει το λόγο. Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Χαίρομαι που ξαναβλέπω εδώ τον Πρωθυπουργό της Λετωνίας, που γνωρίζει πολύ καλά το ημικύκλιο γιατί ήταν ευρωβουλευτής για εννέα έτη. Τον χαίρο, χαίρο ιδιαίτερα που τον βλέπω γιατί θυμάμαι πάντα την λετονική προεδρία του Συμβουλίου των Υπουργών και θυμάμαι την προεδρία γιατί ήταν η πρώτη πραγματική προεδρία επί επιτροπής μας. Συνυπάρξαμε για δύο μήνες με την Ιταλική Προεδρία. Θυμάμαι την τελευταία μέρα της προεδρίας αυτής της Λετωνίας. 29 προς 30 Ιουνίου νύχτα υιοθετήθηκε η οδηγία για τα roaming, για τα τέλη περιαγωγής, εξασφαλίζοντας την ελεύθερη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στην τηλεφωνία και το ίντερνετ. Κάτι που αποδεικνύει ότι η Ευρώπη μπορεί να πετύχει και πρέπει να κρατάμε την ελπίδα μας μέχρι τελευταία μέρα συχνά συζητούμε, σαν να μην είχαμε άλλο πράγμα να κάνουμε για το Brexit. Πριν τι εκλογέ θα ήταν, θα ίσως σκόπιμο να τονίσουμε προς τους πολίτες τι επιδόσεις της Ένωση τα τελευταία χρόνια. ιδίω την χρήσιμη απόφαση για την περιαγωγή. Σημαντικό είναι το Brexit, σημαντικότερη η καθημερινότητα των πολιτών. θελήσαμε να είμαστε και γίναμε η Επιτροπή του Διαλόγου. Οργανώσαμε συναντήσεις με τους πολίτες. 1.600 συναντήσεις διαλόγου με τους πολίτες. Κάτι που αποδεικνύει ότι οι επίτροποι δεν κλείνονται στα μπούνκερ του και κυκλοφορούν ανά την Ευρώπη. Αυτό αποδεικνύει ότι η Επιτροπή δεν είναι μια συμμορία πραξικομα χωρίς νομιμοποίηση, αλλά είμαστε σε καθημερινή επαφή με τους πολίτες. Η Ευρώπη δεν μπορεί να γίνει χωρίς να το θέλουν οι πολίτες, χωρίς τα έθνη. Τα έθνη είναι σημαντικά. Αυτοί που πιστεύουν ότι τα έθνη είναι μια προσωρινή δημιουργία της ιστορίας, σφάλουν. Οι, τα έθνη έχουν διάρκεια δεν πρέπει λοιπόν να μιλάμε για Ηνωμένε Πολιτείε τη Ευρώπης πλέον, διότι δίνει την εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται κράτος. Η Ευρώπη δεν θα γίνει ποτέ ένα κράτος που θα αντιγράψει το μοντέλο των Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης. Είστε Λετωνός, Βαβαρός, Βρετόνος, Γάλλος, Λουξεμβουριέζος και Ευρωπαίος. Δεν υπάρχουν αντιβάσεις στον πατριωτισμό αν ο πατριωτισμός είναι υπεύθυνο και αντιλαμβάνεσαι την ανάγκη, την συμμετοχή σε ένα ευρύτερο σύνολο που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς ως Επιτροπή θελήσαμε να πάψουμε να παρεμβαίνουμε σε όλα τα μικρά γεγονότα της καθημερινότητας των πολιτών και να στραφούμε στα μεγάλα ζητήματα που διακυβεύονταν στο μέλλον. Αυτό ήταν και η συμφωνία που είχαμε κάνει μαζί σας, τους εκπροσώπους των λαών της Ευρώπης όταν το καλοκαίρι του 2014 είχα υποβάλει τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές της πολιτικής της Επιτροπής μας. Δεν ήταν ε, λόγια του αέρα. Είχαμε υποβάλει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που προωθήσαμε ήδη την πρώτη χρονιά. Μέχρι σήμερα. 350 από τις προτάσεις μας έχουν εγκριθεί ενώ 164 παραμένουν ακόμα στην τράπεζα του, στο τραπέζι των συνομοθετών. Εγώ θα είχα βέβαια ε, την επιθυμία να προχωρήσουν όλες οι μεταρρυθμίσεις που είχαμε προτείνει για το καθεστώς του ασύλου, για παράδειγμα. Ωστόσο, πρέπει να πω ότι ποτέ δεν είχαμε τόση πολύ πρόοδο στα κοινωνικά ζητήματα που για πολλά χρόνια ήταν ο φτωχός συγγενής της ανάπτυξης της Ευρώπης. Αυτό θα έπρεπε να... Αυτό άλλαξε και, προ... τώρα η, προσπάθεια του, της Επιτροπής είναι ακριβώς να συνοδεύονται οι δύο κατηγορίες. Η Λετωνία είναι μια χώρα που αξίζει και άξιζε την συμμετοχή της στην Ένωση, όπως τόνισε και ο Πρωθυπουργό της Λετωνίας πριν από λίγο λόγια. Είχα, είπατε, ε, κύριε Πρωθυπουργέ, ότι όντως η χώρα σας ανέλαβε τις ευθύνες της και πραγματικά όπως λένε οι ποιητέ σας, ε, θα, θα, θα είμαστε τόσο μεγάλοι όσο μπορούμε, όσοι θέλουμε να είμαστε. Και αυτό το πετύχατε. Αγωνιστήκατε για την ελευθερία σας κάτω από πολύ πιο δύσκολες συνθήκες από αυτές που φαντάζονταν οι Δυτικοευρωπαίοι. Κάνατε ιστορία αντί να υποστείτε πίεση από τους μεγάλους, όταν υποστήκατε τις πιέσεις από τους μεγάλους γείτονές σας. Είπατε όχι στα όπλα. Επιδιώξατε με ειρηνικό τρόπο την ελευθερία σας. Και αποτελείτε, και αυτό αποτελεί ένα από τα καλύτερα συμβάντα της σύγχρονης ιστορίας. Ο τρόπο με το οποίο η Λετωνία και οι άλλες βαλτικές χώρες αγωνίστηκαν για την ανεξαρτησία τους. Η Λετωνία δεν έχει θέση στο σκοτάδι, στη σκιά, αλλά στον ήλιο, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πραγματικά μια μεγάλη μέρα η μέρα στην οποία η Λετωνία έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπήκαμε στην, ε, μπήκατε στην, ε, στο Σέγγεν και σύμφωνο απόλυτα με αυτά που είπατε για τα ιστορικά σύνορα και την, ε, τα ιστορικά σύνορα. Την ασφάλεια αυτών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ακτοφυλακή, συνοριοφυλακή με 10.000 ε, προσωπικό, άντρες και γυναίκες. Το Συμβούλιο ήθελε να αναβάλει την πρόταση αυτή για το 2027. Ζητήσαμε εμείς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2020. Όλοι όμως λένε ότι πρέπει να προστατεύσουμε τα εξωτερικά μας σύνορα. Ας το κάνουμε λοιπόν πραγματικότητα. βοηθάτε να καταστεί η Ευρώπη πιο δυνατή και πιο ασφαλής. Είσαστε ένα από τα 25 κράτη-μέλη που ξεκίνησε την συνεργασία στα θέματα άμυνας τον Δεκέμβριο του 2017 και χαίρομαι που διαδραματίζεται σημαντικό ρόλο και σε άλλα σημαντικά θέματα σε ό,τι αφορά την στρατιωτική κινητικότητα και τη διευκόλυνση αυτής. Είναι σημαντικό αυτό για τη Λετωνία, η στρατιωτική κινητικότητα. Καθιστάτε λοιπόν ε, την κινητικότητα αυτή πιο εύκολη και κοιτάξτε, κοιτάξτε και το θέμα των ε, ζητημάτων αυτών και το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση επηρεάζει και ενισχύει την ενεργειακή επικυριαρχία και την εθνική επικυριαρχία. Κοιτάξτε τα θέματα ενέργειας, για παράδειγμα, που αποτελούν σημαντικό τμήμα της ευρωπαϊκής πολιτικής, την ιστορία σας και τη γεωγραφία σας, που σημαίνουν ότι η Λετωνία και η Βαλτική ήταν αποκομμένοι από την υπόλοιπη Ευρώπη. Αναλάβαμε τα καθήκοντά μας λοιπόν και τότε ξεκαθαρίσαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα αφήσει σε καμία περίπτωση τους πολίτες της να κρυώνουν και στο σκοτάδι. Για μένα αυτό τότε ήταν θέμα της Βαλτικής, ναι, αλλά όχι μόνο θέμα της Βαλτικής, αλλά ήταν και ευρωπαϊκό ζήτημα. Και γι' αυτό λοιπόν όταν αλάβαμε τα καθήκοντά μας ιδρύσαμε μια ενεργειακή ένωση και τη βάλαμε στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας για να μπορέσει και η Βαλτική και η Λετωνία και οι υπόλοιπε βαλτικές χώρες να δουν ότι οι ενεργειακέ του ανάγκε καλύπτονται. Σήμερα λοιπόν εξυγχρονίζουμε την αγορά του ηλεκτρισμού. Μέχρι το 2025 επενδύουμε σε υποδομές και έχουμε την πιο φιλόδοξη πολιτική σε όλο τον κόσμο σε ό,τι αφορά την ενέργεια και το κλίμα. Είμαι ευτυχής που αυτή η αυτό το όραμα της Ενεργειακής Ένωσης υλοποιήθηκε και κατέστη πραγματικότητα και ευχαριστώ τον Πρωθυπουργό για την ηγεσία του και για τη δουλειά που έκανε ως Πρωθυπουργό σήμερα και ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο παρελθόν. Κύριε Πρόεδρε, αλλάζω γλώσσα. Η Λετωνία συμβάλλει στην Ευρώπη. Αυτό θεωρώ ότι είναι φυσιολογικό και γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι είναι φυσιολογικό και η Ευρώπη να επενδύσει στην Λετωνία γιατί επένδυση στη Λετωνία είναι επένδυση στο ευρωπαϊκό μέλλον. Οι Λετωνοί γνωρίζουν από πρώτη χέρι τι αντίκτυπο μπορεί να έχει αυτό. 50.000 ε, Λετωνοί αναζητούν ε, δουλειά από το 2014 στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αναζητούν επίση νέε δεξιότητε, νέε ικανότητε για να μπορέσουν να απορροφηθούν από την αγορά εργασία. 300 χιλιόμετρα νέα κτίρια και νέοι δρόμοι χρηματοδοτήθηκαν από ευρωπαϊκού πόρου για να συνδέσουν και, τις, ε, και να αναπτύξουν και τις ε, αστικές περιοχές αλλά και την Ήπεθρο στη Λετωνία. 960 δισεκατομμύρια επενδύσεις στη Λετωνία κινητοποιήθηκαν. Το μέλλον της Λετωνίας λοιπόν αφορά όλους μας, είναι το μέλλον όλων μας και γι' αυτό λοιπόν προτείνουμε στον επόμενο προϋπολογισμό 100 δισεκατομμύρια ευρώ στην καινοτομία και στην έρευνα να επενδυθούν. Θέλουμε να επενδύσουμε στο μέλλον της Ευρώπης γιατί μόνο από κοινού και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του μέλλοντος. Για παράδειγμα, θα τριπλασιαστούν ε, οι επενδύσεις στην ασφάλεια και θέλουμε επίσης και στο θέμα να υποστηρίξουμε τα, τους πόρους και τις επενδύσεις για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, το Erasmus Plus. Διπλασιάζονται οι πόροι μάλιστα για το πρόγραμμα αυτό. Ευχαριστώ τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνησή του για την διαρκή υποστήριξη και την ενεργή συμμετοχή του. Να κάνω κάποιες ε, παρατηρήσεις όμω και σε ό,τι αφορά τις μεσοπρόθεσμε επενδύσεις και τον προγραμματισμό. Όντω. στην έρευνα, στην ανάπτυξη, στην εκπαίδευση, στην νεολαία επενδύουμε. Όλα αυτά όμως μπορούμε να τα κάνουμε μόνο αν γίνουν περικοπέ σε άλλες πολιτικές, συνοχή και σε γεωργία. Αυτό δεν με ικανοποιεί σε καμία περίπτωση, αλλά αν αφήσουμε τα πράγματα όπως έχουμε και προσθέσουμε και τι νέε προτεραιότητες, καπάκι, επί των οποίων συμφωνήσαμε, πολύ απλά θα καταρρεύσει ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός στο επίπεδο του 1,4%. Αυτό το θέλει κανεί. Εμένα δεν θα με ενοχλούσε καθόλου, ξέρετε, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση αξίζει παραπάνω από 1,4% του ΑΕΠ της. Αλλά ακόμα και το ίδιο το Κοινοβούλιο σε θέματα δημοσιονομικά είναι λιγότερο διστακτικό μεν από το Συμβούλιο, αλλά ω ανώτατο όριο για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό έφτασε το 1,3%. Αν εμείς ε, από Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προτείνουμε 1,4%. Ούτε ακόμα και εσείς στο Κοινοβούλιο δεν θα συμφωνούσατε με το 1,4%. η γεωργία και η συνοχή είναι πολύ σημαντική τομείς και για κάποιες χώρες πιο σημαντική από ό,τι για άλλες βέβαια. Η Λετωνία έχει σημαντικά χρόνια, σημαντικό παρελθόν, όχι μόνο λόγω της γεωγραφικής ε, της θέσης, αλλά και της ε, ιστορίας της, αλλά και λόγω των οικονομικών κρίσεων που έπληξαν την Λετωνία. Πέντε χρόνια ωστόσο μετά την ε, έναρξη της αντιμετώπισης της κρίσης η Λετωνία τα πηγαίνει καλύτερα. Και αυτό αποτελεί και επίτευγμα του προκάτοχου σας, του κυρίου Βαλτίς Ντομπρόφσκι, του προκατόχου σας, ο οποίος έθεσε στη σωστή πορεία τη Λετωνία. Και γι' αυτό κατέβαλα ιδιαίτερες προσπάθειες ε, να καταστεί εκ νέου επίτροπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιος για θέματα νομισματικά. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαλντής. Πολλά λοιπόν θα είχα να πω για αυτά που μας παρουσίασες. Μίλησες πάρα πολύ ώρα όμως και έτσι αναγκαστικά εγώ θα πρέπει να κλείσω σιγά σιγά. Η Λετωνία είναι μικρή χώρα και εγώ είμαι ειδικό στις μικρές χώρες, ξέρετε. Είναι όμως μια χώρα με μεγάλες φιλοδοξίες. Είναι το μέρος όπου συναντιέται η Ανατολή με τη Δύση. Δεν μπορεί η Ανατολή και η Δύση να διχάζονται. Είναι οι δύο πνεύμονες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αν η Ευρώπη θέλει να έχει ένα καλό ε, μέλλον, θα πρέπει να αναπνέει και με τους δύο πνεύμονες της. Είναι η τελευταία αυτή ομιλία που απευθύνω προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με βαριά καρδιά. Βλέπω ότι μερικοί συνάδελφοι αποχωρούν από την πολιτική και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρέπει να σας πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ η δουλειά εδώ στους κόλπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έμαθα πολλά, τσακώθηκα πολύ, αλλά θεωρώ ότι πετύχαμε και πολλά. Είχα πει την πρώτη μέρα της ε, των καθηκόντων μου η Ευρώπη είναι κάτι το οποίο πρέπει να ζήσει κανείς. Αν δεν τη ζήσουμε, δεν ζει η αγάπη μας ε, αυτή για την Ευρώπη. Εγώ αγαπώ την Ευρώπη και ε, μακάρι να ζήσει καλά η Ευρώπη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε της ε, Κομισιόν, αγαπητέ Ζων Κλοντ. Ευχαριστώ πολύ για την συνεργασία μας, παρόλο ότι μερικές φορές είχαμε και κάποιες πιο... Ε, είχαμε μερικές στιγμές έντασης στις συζητήσεις μεταξύ της Κομισιόν και του Κοινοβουλίου. Για τα πιο σημαντικά όμως θέματα ε, εργαστήκαμε μαζί προς όφελος και προς συμφέρον των πολιτών μας, των Ευρωπαίων πολιτών. Έχουμε ανάγκη την Ευρώπη. Προφανώς χρειάζεται να τη βελτιώσουμε, να την αλλάξουμε. Αλλά είναι ο μόνος τρόπος ε, έτσι ώστε η Ευρώπη να προστατεύσει, να υπεραμυθεί της Ευρώπης και να προστατεύσει τους πολίτες της. Θυμάστε τι έγινε πριν μερικέ μέρες στην Παναγία των Παρισίων. Ε, η, η γενικευμένη θλίψη που προέκυψε απέδειξε ότι έχουμε μια κοινή ψυχή, μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες παρόλο που μπορεί να μιλάμε διαφορετικές γλώσσες. Ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν για το έργο σου, για την προσήλωσή σου, για το πάθος σου και θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε. Θα τα ξαναπούμε στο Συμβούλιο βέβαια. Ε, αλλά χαίρομαι που ήσουν εδώ σήμερα και όλες τις προηγούμενες φορές. Συγχαρητήρια. Πρέπει να κλείσουμε ε, την εγγραφή για το Catch the Eye. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Βέμπερ. Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, κύριε Πρωθυπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, πολύ σπουδαία ομιλία και να ευχαριστήσω τον ε, Πρόεδρό μας που διοργάνωσε αυτή την ομιλία στα πλαίσια του μέλλοντο τη Ευρώπη και χαιρόμαστε που Κριστιανή είσαι εδώ μαζί μα, ω τελευταίο ομιλητή εδώ στην Ολομέλεια μεγάλη η συμβολή σου και η παρέμβασή σου για το μέλλον της Ευρώπης και όλοι έχουμε την αίσθηση ότι βλέπουμε πώς μιλάει η Ευρώπη, πώς μιλάει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα ήταν καλό στο μέλλον να έχουμε πιο πολλούς πρωθυπουργού πρώην μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αυτό πραγματικά το απολαύσαμε σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και αυτό πραγματικά που μου άρεσε είναι ότι ξεκινήσατε με αισιόδοξο μήνυμα. Μιλάμε για το μέλλον της Ευρώπης, μιλάμε για τη χώρα σας, τη Λετωνία, μια επιτυχής ιστορία τις τελευταία χρόνια και με την υποστήριξη του κυρίου Ντομπρόφσκη ε, υπό την ηγεσία του μεγάλη οικονομικέ ε, επιτυχίε, μεγάλη επιτυχία για τη χώρα σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις τις οποίες ανέφερε ο Ζαν Κλοντ Ιούνκερ και για το αίσθημα της ασφάλειας, ότι οι Ευρωπαίοι αισθάνονται ασφαλείς και προστατευμένοι, γιατί αυτό είναι τμήμα μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ό,τι αφορά και τη Ρωσία και τι εξωτερικέ ε, απειλέ. Είναι επιτυχημένη ιστορία γιατί μιλάμε για την ε, εντολή που μας έχει δοθεί. Αυτό το αναφέρει και ο κύριος Γιούγκα. Ανέφερε το ότι επιτύχαμε στο θέμα της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων εκατομμύρια νέων θέσεων απασχόλησης ε, που συστήθηκαν με το πρόγραμμα Γιούγκα, η βιώσιμη ανάπτυξη και η κορονίδα ήταν ε, ο αγώνας κατά της κλιματικής αλλαγής. Άρα δηλαδή μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι και ευχαριστημένοι για όλα αυτά που καταφέραμε από την καθοδήγηση του κυρίου Γιούγκα. Και κάτι άλλο. Εγώ είμαι 46 ετών. Είμαι, ε, ανήκω σε αυτή την γενιά που μπορεί να πει ότι έζησε εν ειρήνη η προηγούμενη γενιά, ε, ναι, είχε και αυτή ειρήνη, αλλά είχαμε το σιδηρούν παραπέτασμα και η προπροηγούμενη γενιά είχε πόλεμο. Αυτό λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, πρέπει να το έχετε κατά νου όταν θα κάνετε την προεκλογική σας εκστρατεία. Είναι πολύ σημαντικό σήμερα το να ζούμε στην Ευρώπη και θα προστατεύσουμε την Ευρώπη από όλους τους ε, εθνικιστές και τους εγωιστές. Το δεύτερο θέμα που αναφέρατε είναι εκείνο που είναι πολύ συγκεκριμένο, οι απαντήσεις στις ερωτήσεις, στις ανησυχίες των ανθρώπων. Αναφέρατε τη μετανάστευση. Συμφωνούμε απόλυτα με αυτά που είπατε για την προστασία των συνόρων μας. Ε, ε, Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα πρόγραμμα μετεγκατάστασης, ένα ε, φιλόδοξο πρόγραμμα και χρειαζόμαστε και ένα πρόγραμμα για την Αφρική. Ίσως στο μέλλον να έχουμε και έναν επίτροπο για την Αφρική που θα συνδυάζει όλα αυτά που χρειαζόμαστε για την Ήπειρο αυτή. Ε, ξάλλου, τα περιφερειακά ταμεία είναι καθοριστική σημασία. Ε, το εμπόριο είναι καθοριστική σημασία και η κοινή αγορά. Πρέπει να ενισχυθεί η κοινή αγορά γιατί Καταρχήν, πρώτα απ' όλα πρέπει εδώ να δημιουργήσουμε θέσει απασχόληση. Και τέλο και η κλιματική αλλαγή, όλα αυτά υπάρχουν στο θεματολόγιο, αλλά όταν μιλάμε για το μέλλον τη Ευρώπη πρέπει να είμαστε και ειλικρινεί. Γιατί υπάρχει ένα πράγμα που είναι απόλυτα σαφέ. εντάξει είναι η πολιτική προσέγγιση, αλλά το άλλο σημαντικό θέμα είναι η μέθοδο. Πώ θα επιτύχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Και εκεί υπάρχουν προβλήματα. Χρειαζόμαστε μια ισχυρότερη Ευρώπη, αλλά υπάρχει το πρόβλημα τη ομοφωνία. Εγώ το αποκαλώ πρόβλημα την ομοφωνία. Γιατί α πούμε όταν πρόκειται για τη Ρωσία πρέπει και 27 χώρε να συμφωνήσουν. Γι' αυτό πρέπει να αρθεί η ομοφωνία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να γίνει ένα ισχυρό πολιτικό παίκτη ε, με παγκόσμια και ε, ουσιαστική εμβέλεια. Άρα πρέπει να γίνουν κάποιε αλλαγέ. Και όταν μιλάμε για μεθόδου, ε, νομίζω ότι πρέπει να ξεπεράσουμε αυτή τη μέθοδο τη έγερση γεφυρών. Α αναφερθούμε στη δική μου τη χώρα, η Γερμανία η Γερμανία ήταν ε, κατά της άποψης ε, του να υπάρχει υπάρχουν συγκεκριμένες ποσοστώσεις ε, για την ε, κατανομή των μεταναστών μέχρι το 2015. Το 2015 να γιατί, γιατί τότε εμφανίστηκε το πρόγραμμα στη Γερμανία και μέσα σε τρει μόνο μήνε η Γερμανία άλλαξε γνώμη και ζήτησε ένα δεσμευτικό μηχανισμό ποσοστώσεων στην Ευρώπη. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν πρέπει κανεί να εξετάζει τα προβλήματα τη Ευρώπη κάτω από εγωιστικό πρίσμα. Πρέπει να μάθουμε να έχουμε κατά νου και τη θέση των υπολείπων και των άλλων όταν, εάν μάλλον θέλουμε μια ισχυρή Ευρώπη. Και τέλος ένα μήνυμα, ε, μια Ευρώπη δημοκρατική. Γνωρίζετε για τι πράγμα μιλάμε. Είναι θέμα δικαιώματος ανάληψης ε, πρωτοβουλίας. Το να μπορεί το Κοινοβούλιο να διεξάγει περισσότερες έρευνες, να εξετάζει και το Κοινοβούλιο την εφαρμογή των κανόνων και χαίρομαι πάρα πολύ κύριε Πρωθυπουργέ που στηρίζει την ιδέα του Spitzenkandidat, του βασικού εκπροσώπου μιας πολιτικής ομάδας. Εγώ παραδείγματο χάρη είμαι Spitzenkandidat και ζητώ την υποστήριξή σας. Και τέλος μέλλον της Ευρώπης σημαίνει ότι πρέπει να προστατεύσουμε την πεμπτουσία της Ευρώπης. Μιλήσαμε για δημοκρατικό τρόπο ζωής, αλλά δημοκρατία ανεξάρτητη από τη δικαιοσύνη ή συμμεταχείριση όλων των ανθρώπων και δικαίωμα στην ελευθερία έκφραση, στην ελευθερία του τύπου. Όλα αυτά τα δικαιώματα πρέπει να τα εγγυηθούμε στο μέλλον, να υπάρχει ο απαραίτητο μηχανισμό. Να δώσουμε στον κόσμο ε, το καλό πρότυπο, το καλό παράδειγμα, πώ μπορεί κανεί ε, να ζει σε μια δημοκρατική Ευρώπη με ανθρώπινο τρόπο. Ο δημοκρατικό τρόπο ζωή είναι μια προσφορά στην Ευρώπη και αυτό ακριβώ είναι το μέλλον τη Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πολύ. Και... τώρα για τους σοσιαλιστές η κυρία Μπρέσο παρακαλώ. Κύριε Πρωθυπουργέ, είναι μεγάλη τιμή σήμερα να σας καλωσορίσω, καθώς έχετε αναλάβει τα νέα σας καθήκοντα ως Πρωθυπουργός σε αυτό το ημικύκλιο. Και εσείς φυσικά το γνωρίζετε καλά, γιατί ήσασταν Ευρωβουλευτής περίπου για 10 χρόνια. Και είναι ακόμα μεγαλύτερη τιμή γιατί εσείς είστε όχι μόνο ο τελευταίος αρχηγός κυβέρνησης πριν από τις επόμενες ευρωεκλογέ, αλλά επειδή στην ομιλία σας αναφέρατε σημαντικές προοπτικές για την Ένωση που θα έχουμε το καθήκον να οικοδομήσουμε μετά τις 26 Μαΐου. Και γι' αυτό τον λόγο σας καλωσορίζουμε εκ μέρου των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών ω τελευταίο αρχηγό κυβέρνηση που έρχεστε να επισκεφτείτε το Κοινοβούλιο με τι εκλογέ. Η επίσκεψη σα αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία για να συζητήσουμε για τη χώρα σας, τη Λετωνία και το ρόλο της εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για μα, ε, τους ευρωβουλευτές, είναι πάντοτε κάτι θετικό να συναντάμε έναν από τους ε, πρώην συναδέλφου μας ε, να εκπροσωπούν μια εθνική κυβέρνηση και ελπίζουμε να αυξηθούν οι συνάδελφοι. Εδώ θέλουμε να εκφράσουμε μια συγκεκριμένη φιλοδοξία των Ευρωπαίων πολιτών, να οικοδομήσουμε μαζί μια ισχυρή ένωση για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του καιρού μας. Μένει μόνο ένα κράτος μέλος, είτε πρόκειται για ένα μικρό κράτος όπως το δικό σας, είτε για μια μεγαλύτερη χώρα όπως η Ιταλία ή η Γαλλία ε, δεν ε, μπορεί κανένας να κάνει μόνος του τίποτα για να καταπολεμήσει την κλιματική αλλαγή, ούτε να ε, διασφαλίσει τη δική του άμυνα ή την οικονομική ανάπτυξη της χώρας του. Κύριε Γιούνκερ, όπως και εσείς και εγώ αγαπώ την Ευρώπη, αλλά αγωνίζομαι για τα ενωμένα ευρωπαϊκά κράτη, στον πληθυντικό. Και επομένως ε, δεν βλέπω που είναι το πρόβλημα. Σας ευχαριστούμε πάντως για τη δεσμευσή σας για την Ευρώπη και από την πλευρά της δικής μας ομάδας ε, καθώς ε, είναι η τελευταία παρουσία σας στο Κοινοβούλιο σήμερα, όπως είπατε. Εμείς ε, έχουμε εκτιμήσει τη δέσμευσή σας για μια Ενωμένη Ευρώπη που ίσως να πηγαίνει πιο πέρα από τα Ενωμένα ΕΕ κράτη της ε, Ευρώπης. Ελπίζουμε όσα είπατε να αποτελούν μια μεγαλύτερη ευρωπαϊκή δέσμευση της κυβερνήσή σας, ε, κύριε Πρωθυπουργέ, που μέχρι τώρα έχει δείξει κάποια αμφίσιμα σημεία σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊστικό σας χρώμα. Σε ένα πλαίσιο όπου τα μεμονωμένα κράτη δεν μπορούν να παίξουν ρόλο στη διεθνή σκηνή, θα, μήπως ε, θα έπρεπε να θέσουμε τέλος τον κανόνα ομοφωνίας ε, στο Συμβούλιο που κι εσείς υποστηρίζετε. Ο κανόνας αυτός προωθεί μόνο τα μεμονωμένα συμφέροντα των κρατών μελών εις βάρος του γενικού συμφέροντος της Ένωσης. Θέλετε να συνεχίσετε να ε, αποτελείτε το φύλακα ενός κονκλαβίου όπου οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται ή συχνά αναβάλλονται η παρουσία μιας ισχυρής Ευρώπης είναι κάτι απαραίτητο και το υπενθυμίσατε. Ε, θα πρέπει να δείτε πού θέλετε να βρεθείτε στα βιβλία τη ιστορία από την πλευρά του συμφέροντο των Ευρωπαίων πολιτών ή στην πλευρά όσων έχουν υποστηρίξει το συμφέρον ε, κάποιων ελίτ. Και θέλω να επιμείνω. Θέλετε να βρεθείτε στην πλευρά όποιων ε, κατέστησαν ένα κατέστησαν αδρανές το ευρωπαϊκό οικοδόμημα ή από την πλευρά όσους έδωσαν στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα τα χρήσιμα εργαλεία προκειμένου να αναπτύξει τη δυναμική δική του. Για μας, για του σοσιαλιστέ και δημοκράτε, η Ευρώπη οικοδομείται μέσω του νόμου και με σεβασμό φυσικά, ε, σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, αλλά και των δικαιωμάτων των πολιτών. Από τον Ιανουάριο ε, κάποιες δηλώσεις που κάνετε έχουν προκαλέσει πολλές ερωτήσεις και θέλουμε απαντήσεις σε σχέση με την ευρωπαϊκή δέσμευση για την μετεγκατάσταση των προσφύγων στην Ευρωπαϊκή. Εσεί είπατε ότι είστε κατά. Όμως, πώς ε, θα γίνει αυτή η ανακατανομή ε, όταν ε, έχουμε κοινά σύνορα. Η θέση αυτή έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της ελεγγύης που εφαρμόζεται σε όλες τις κοινοτικέ μας πολιτικές, παραδείγματο χάρη και στην πολιτική συνοχή. Τι μπορείτε να μα πείτε λοιπόν συγκεκριμένα για αυτό το ζήτημα. Τώρα, τι λέτε για την έρνησή σας να υποστηρίξετε την έρεξη σε υπερβάσιβα του άρθρου 7 κατά Πολωνίας και Ουγγαρίας. Πώς εξηγείτε αυτή την έρνησή σας με τις σωστές επικρίσεις στην πολιτική του Πούτιν και την υποστήριξή σας σε κάποια μέρη ε, της ε, ε, δεξιάς από το Σολβίνι στον Όρμπαν τώρα. Δεν θεωρείτε λοιπόν ότι αυτό αποτελεί αντίφαση και τελευταίο σημείο, αλλά σημαντικό ποια είναι τα μέτρα που έθεσε εφαρμογή η κυβέρνησή σας σε σχέση με την όξυνση των διακρίσεων απέναντι στους λοάδμα. Ε, στην ανακοίνωση Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του ρατσισμού, αυτή η Επιτροπή δείχνει πολύ μεγάλες τις λειτουργίες σε ό,τι αφορά την υλοποίηση μέτρων για την προστασία των μειονοτήτων. Η Ένωση μας προωθεί ε, την ε, ανοχή και ε, εσείς θα πρέπει να σέβεστε τις αξίες. Σας ευχαριστώ Κνέου, για την ομιλία σας και για τις απαντήσεις που θα δώσετε στις ερωτήσει μου. Ευχαριστώ. Τώρα το ρόλο έχει ο κύριο Τσίλα από το ECR. Πρόεδρε, Χαίρομαι πάρα πολύ κύριε Πρωθυπουργέ που σας έχουμε εδώ και που άκουσα το τόσο όμορφο περιεχόμενο της ομιλίας σας. Θα ήταν πολύ καλό να δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό. Θέλω τώρα να επιστήσω την προσοχή σας και στις κυρίες που συνοδεύουν τον ε, κύριο Κάρινς. Μπορούμε να είμαστε πραγματικά περήφανοι για αυτές. Είναι γυναίκες της διπλωματίας και πράγματι είμαστε περήφανες για αυτές. Θυμάμαι την ημέρα που ενταχθήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη. Πολλές φορές όμως έχω λυπηθεί για διάφορες πτυχές της ευρωπαϊκής πολιτικής, όπως επίσης και για την εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν είναι τόσο καλή. Και γι' αυτό ακριβώς θέλω να μιλήσω. Η ομιλία σας δεν είπε ότι όλα είναι ωραία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ας συνεχίσουμε ειρηνικά να εκτιμούμε τα επιτεύγματά μας και να φροντίσουμε για μια ακόμα πιο ενωμένη Ευρώπη. Χαίρομαι που βάλατε αποχρώσεις αυτό. Το ECR ήταν πάντα η πολιτική οικογένεια η οποία υποστήριζε την πραγματική ενιαία αγορά σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Και ξέρω ότι έχετε κι εσείς κάποιες αμφιβολίες. Είπατε ότι δεν χαίρεστε πάρα πολύ με τους Ευρωπαίους ε, πρωταθλητές. Οι εθνικοί πρωταθλητές ίσως να είναι κάτι καλύτερο. Έχουμε διαφωνήσει και με τον κύριο Βέμπερ που λέει ότι θέλει να αλλάξει κάποιες αρχές που διέπουν τις κρατικές επιχορηγήσεις. Νομίζω ότι είναι ένα λάθος μήνυμα προς την οικονομία. Γιατί ωραία, ωραίο το μήνυμα η Ευρώπη που προστατεύει, αλλά που προστατεύει από ποιον, από τον έξω κόσμο. Εντάξει, αλλά τελικά μήπω είναι αυτός ο λάθος δρόμος, μήπω οι περισσότεροι κίνδυνοι υπάρχουν μέσα στην εσωτερική αγορά. Και εδώ μπορώ να σας δώσω παράδειγμα στο οποίο αναφερθήκατε λίγο πολύ κι εσείς που είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε για τα μηδενικά τέλη με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Πρόσφατα εγκρίναμε το πακέτο κινητικότητας. Πολύ επίμαχο θέμα. Και είναι σαφές ότι πολύ ωραία πολλές κυβερνήσεις βαλτικές και από διάφορες πολιτικές οικογένειες ήταν κατά. Οπότε τελικά είναι να αναρωτιόμαστε αν είναι κάτι κακό για τις χώρες της Ευρώπης, είναι δυνατόν να είναι καλό για την Ευρώπη την ίδια. Και αν η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε το ίδιο πακέτο κινητικότητας ε, για τις εμπορικές μεταφορές στις Ηνωμένε Πολιτείε, ώστε να μπορεί κανείς με τον ίδιο τρόπο να κυκλοφορεί από τη Νέα Υόρκη στο Wyoming, θα ήταν καταστροφικό αυτό. Εμείς εδώ μιλάμε για το 1% του ΑΕΠ και ξεχνάμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση το αντίστοιχο είναι το 20% του Αμερικανικού ΑΕΠ. Νομίζω ότι αυτά πρέπει να τα πούμε. Και αν θέλουμε να δημιουργήσουμε μια περισσότερη φεντεριλιστική Ευρώπη, κάτι το οποίο δεν θέλει βέβαια το ΙΣΙΑ, το θέλουν άλλες πολιτικές ομάδες. Έχει καταφέρει πολλά η Λετωνία στην νομοθεσία της για τους μετόχους, για παράδειγμα. Στο Tax 3 δεν αναφέρθηκε όμως και δεν αναφέρονται ε, σαν κακά παραδείγματα άλλες ε, χώρες που δεν βρίσκονται και πολύ μακριά από εδώ από το Στρασβούργο. Έπειτα η έρευνα και η τεχνολογία. Φυσικά και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και φαίνεται αυτό από το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Εσεί το είπατε, αλλά πώ γίνεται η κατανομή. Δημογραφικά θα συνεχίσουμε ακόμα και με ένα ευρύτερο πρόγραμμα, το Horizon, α πούμε, που είναι ένα καλό πρόγραμμα, δεν λαμβάνουμε υπόψη μας τις δημογραφικές αλλαγές στην Ευρώπη που οι διαφορές οι δημογραφικές θα ενισχυθούν στο μέλλον. Αλλιώς θα είναι το δημογραφικό στις περιφερειακές χώρες όπου θα υπάρχουν μεγάλα προβλήματα και αλλιώς θα είναι η κατάσταση στο κέντρο ή στο νότο. Θα υπάρξουν διαφορές ακόμα μεγαλύτερες από ό,τι έχουμε τώρα. Οπότε σε πολλά συμφωνώ μαζί σας, σε πολλά θέλω να πάω ακόμα πιο μακριά. Ελπίζω το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει μια δικιά μας μεγάλη πολιτική οικογένεια ώστε να μπορέσει να ενισχύσει την ενή αγορά που είναι και βασικά ο πυρήνας της Ευρώπης και που θέλουμε να αναπτυχθεί περισσότερο στο μέλλον. Ευχαριστούμε εκ μέρους των φιλελεύθερων ο κύριος Στελίτσκα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ. Σας καλωσορίζουμε και πάλι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κύριε Πρωθυπουργέ, λοιπόν, ε, καλωσορίσατε και πάλι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Στην αρχή της ομιλίας σας κάνατε ένα σχόλιο ότι μάθατε πάρα πολλά πράγματα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Άρα και εγώ ε, θα κάνω ένα παραλυσμό, ένα ψεύτικο θα έλεγα, γιατί με βάση αυτή την παραδοχή θα ήθελα ο Τσέχος ε, Πρωθυπουργό ε, να είναι μέλος ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τότε θα είχαμε μια τελείως διαφορετική πολιτική της τσεχικής κυβέρνησης για τα ευρωπαϊκά θέματα. Αλλά πέρα από αυτό έχετε ένα πλεονέκτημα. Έχετε γνώση και σωστή τοποθέτηση. Νομίζω ότι αυτά είναι απαραίτητα στοιχεία, αλλιώς δεν μπορεί κανείς να εξελιχθεί. Φοβάμαι όμως ότι όλα αυτά δεν συμβαδίζουν με τον παραλυσμό που έκανα με τον Τσέχο. Ε, Πρωθυπουργό. Αναφέρατε επίση το θέμα των γλωσσών. Είμαι σίγουρο ότι μιλάτε πολλέ γλώσσε ή τουλάχιστον καταλαβαίνετε πολλέ γλώσσε. Δεν νομίζω ότι καταλαβαίνετε τσέχικα, αλλά θέλω να σας πω αυτά που είπατε είναι σαν να διαβάζει κανεί το εκλογικό μανιφέστο του δικού μου του πολιτικού κινήματος και αυτό βέβαια καλό είναι, θετικό, γιατί αυτό σημαίνει ότι ανεξάρτητα από το γεγονό ότι ανήκετε στο ΕΛΚ, εγώ ανήκω στου φιλελεύθερου, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα επί των οποίων μπορούμε και πρέπει να αναζητήσουμε ευρωπαϊκέ λύσει. Μία σειρά θεμάτων επί των οποίων μπορούμε να συμφωνήσουμε και με άλλα κόμματα και νομίζω ότι σε αυτό πρέπει να στοχεύουμε στι επικείμενε εκλογέ. Υπάρχουν λοιπόν αρκετά θέματα επί των οποίων μπορούμε να συμφωνήσουμε και θα επιλέξω κάποια θέματα που θίξατε. Απλουστευμένε ε, λύσεις. Αναφερθήκατε σε εθνικιστές, σε λαϊκιστές. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε τα αίτια αυτού του προβλήματος. Τα αίτια των ανησυχιών και της ανησυχίε εκείνων που κάπου τους χάσαμε σε αυτή τη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης. Αλλά πρέπει να είμαστε και ειλικρινείς και δίκαιοι και να πούμε ότι έχουμε ακόμα δουλειά να κάνουμε. Ότι και στις δικές μας τις πολιτικές οικογένειες, στις δικές μας τις πολιτικές ομάδες και τα κόμματα βρίσκουμε εκείνους που προσφέρουν τις απλουστευμένες ή υπεραπλουστευμένες λύσεις. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ε, δούμε τι ακριβώς γίνεται στο πολιτικό τοπίο. Όσον αφορά άλλα θέματα που θίξατε, μιλήσατε για την εσωτερική αγορά, την κοινή αγορά. Νομίζω ότι εδώ στο Κοινοβούλιο δεν υπάρχει κανείς που να μην πιστεύει ότι η εσωτερική αγορά ε, δεν έχει να παρουσιάσει επιτυχίες, ότι πρέπει να εξελιχθεί περαιτέρω. Πράγματι, μόνο το 35% της εσωτερικής αγοράς είναι ανοιχτό, άρα δηλαδή υπολείπεται ένα 65%. Ε, επίσης, είπατε με απόλυτη σαφήνεια ότι υπάρχει συγκεκριμένο λόγο ε, να ε, πηγαίνει κανείς στι ΗΠΑ να κάνει δουλειές, γιατί εκεί στι ΗΠΑ ε, είναι μια ανοιχτή αγορά. Στι ΗΠΑ μία έγκριση και αδειοδότηση χρειάζεται κανεί. Εδώ, εδώ 28. Γι' αυτό λοιπόν το ερώτημα που τίθεται είναι ότι αν πραγματικά θέλουμε μία σωστή εσωτερική αγορά, πρέπει να έχουμε μία ρυθμιστική αρχή για μία ενωμένη αγορά. Επίσης, ε, κάνατε παραλυσμό με τον αθέμητο ανταγωνισμό από την Κίνα και από αλλού. Και συμφωνώ πάλι μαζί σας, δεν πρέπει να επιβάλλουμε προστατευτισμό, αλλά πρέπει να κατανοήσουμε ότι αν ανοίξουμε τις αγορές, και εγώ με πέρα αυτού, τότε το πλεονέκτημα θα είναι στην πλευρά εκείνων που απατούν και εκείνων που είναι μεγάλοι. Γι' αυτό λοιπόν να μην έχουμε αυτά Θα έχουμε εσωτερική αγορά και ξαφνικά οι νεοσύστατες επιχειρήσεις ε, θα είναι στην διαθέση όπως η Microsoft. Άρα δηλαδή τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι πρέπει να δουλέψουμε στα πρότυπα, στις προδιαγραφές, στην πολιτική ανταγωνισμού. Άρα δηλαδή να έχουμε ένα θεμητό πλαίσιο και το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο να έχουμε το θάρρος και τη βούληση να συστήσουμε μια αμυγός εσωτερική αγορά κατά 100%, όχι μόνο 35%. Εγώ είμαι υπέρ αυτού. Επίσης, μιλήσατε για το θέμα των εξωτερικών συνόρων. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, είναι καθοριστική σημασία στο θέμα, αλλά εκεί εξακολουθούμε να αποτυγχάνουμε. Φοβάμαι λοιπόν, αν δούμε λιγάκι την Τσεχία, εκεί υπάρχουν ε, πολλοί ε, που διστάζουν, δεν έχουν τη βούληση να κατανοήσουν ότι ε, όταν θα έχουμε εσωτερική αγορά και ελεύθερη μετακίνηση, τότε πραγματικά θα μπορούμε να διασφαλίσουμε τα σύνορά μας. Τέλος, όσον αφορά την κλιματική αλλαγή και πάλι, ως προς την κλιματική αλλαγή θα μπορούσαμε να δουλέψουμε σε όλα τα πολιτικά κόμματα και το τελευταίο σημείο ε, θίξατε την κοινή γεωργική πολιτική, την σωστή μεταχείριση των αγροτών. Πράγματι, δεν έχουμε κοινή γεωργική πολιτική γιατί ε, σε πάρα πολλούς εθνικούς ε, προϋπολογισμούς ε, προβλέπονται επιπρόσθετες επιδοτήσεις πέρα από τις προβλεπόμενες. Άρα δηλαδή πρέπει να υπάρχει δίκαιη μεταχείριση των επιχειρηματιών, των καταναλωτών και βεβαίως και των γεωργών. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι θα πρέπει, λέει ο Πρόεδρος, να σεβόμαστε το ο χρόνο που έχει προβλεφτεί για τον κάθε ένα από εσά, έτσι ώστε να υπάρχει και χρόνο για τη διαδικασία Catch the Eye. Εκ μέρου τη αριστερά, ο κύριο Παπαδημούλη. Η σημερινή συζήτηση είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί σε λίγες ώρες ολοκληρώνονται οι εργασίες της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι η τελευταία ομιλία του Προέδρου Γιούνκερ ενώπιον της Ολομέλειας και υποδεχόμαστε τον λετονό πρωθυπουργό ο οποίος ήταν και για εννιά χρόνια συνάδελφός μας στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και είναι ο δωδέκατος πρωθυπουργός που έρχεται εδώ να συζητήσουμε για το μέλλον της ευρώπης σαράντα μέρες πριν τις σημαντικές ευρωεκλογές που έχουμε μπροστά μας. δεν νομίζω ότι είναι η ώρα να αυτοεπαινούμαστε και να επισημαίνουμε τα κάποια θετικά που έχουν γίνει αλλά να δούμε το μέλλον τις προκλήσεις του μέλλοντος και όσα δεν έχουμε κάνει ή όσα έχουμε κάνει λάθος για να καταλάβουμε ότι αυτό είναι ο τρόπος να αντιμετωπίσουμε την ανερχόμενη λαϊκίστικη ακροδεξιά που θέλει να διαλύσει και την ευρωπαϊκή ενοποίηση ως σχέδιο και να διαλύσει τις κοινωνίες μας αναφερθήκατε κύριε κάρινς στον μύθο τον αρχαιοελληνικό του εσώπου με τις βέργες. μία βέργα σπάει εύκολα πολλές βέργες μαζί δεν σπάνε. σωστό. αλλά πρέπει να δούμε εμείς στην ευρωπαϊκή ένωση πού βρισκόμαστε δέκα χρόνια μετά την κρίση της lehman brothers. έχουν μεγαλώσει οι ανισότητες οι κοινωνικές και οι περιφερειακές έχει υποχωρήσει μέσα στην ευρώπη το κράτος δικαίου και η κοινοβουλευτική δημοκρατία το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και η κομισιόν έχουν ζητήσει εναντίον των κυβερνήσεων της πολωνίας και της ουγγαρίας την ενεργοποίηση του άρθρου 7 και στο συμβούλιο δεν κάνετε τίποτα απέναντι στις παραβιάσεις της δημοκρατίας το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και η κομισιόν έχουν ολοκληρώσει μια πρόταση για τη μεταρρύθμιση των πολιτικών ασύλου επτά συνολικά φακέλους και στο συμβούλιο οι κυβερνήσεις δεν κάνετε τίποτα. η κομισιόν η ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα και το ευρωκοινοβούλιο θέλουν την ολοκλήρωση της τραπεζικής ενοποίησης με τον τρίτο πυλώνα που αφορά στο ευρωπαϊκό σύστημα εγγύησης καταθέσεων και στο συμβούλιο δεν κάνετε τίποτα. ακριβέστερα κάποιες κυβερνήσεις όπως της γερμανίας και της ολλανδίας ουσιαστικά έχουν βάλει βέτο. αν θέλουμε λοιπόν να προχωρήσει η ευρώπη και να γίνει πιο ισχυρή η πολιτική ενοποίηση ισχυρότερη η πολιτική διαφάνεια να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή να κάνουμε περισσότερα πράγματα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής όπως μας ζήτησε χθες η 16χρονη γκρέτα Τούμπερκ τότε θα πρέπει να σταματήσει η ευρωπαϊκή ένωση κύριε βέμπερ να είναι μια ομάδα κρατών όπου συζητούν 28 και στο τέλος αποφασίζουν οι γερμανοί. αυτό πρέπει να αλλάξει. και θέλω να σημειώσω ότι συμφωνώ με την παρατήρηση του προέδρου Γιούνκερ ότι για να υπηρετήσουμε τους στόχους που έχουν τεθεί χρειάζεται και ένας ισχυρότερος κοινοτικό προϋπολογισμός με περισσότερα χρήματα στο κοινό ταμείο γιατί πρέπει να μην περικοπούν αλλά αντίθετα να ενισχυθούν τα κονδύλια για την κοινωνική συνοχή. Να μην περικοπούν, αλλά αντίθετα να ενισχυθούν τα κονδύλια για την κοινή αγροτική πολιτική να δώσουμε περισσότερα χρήματα για την νεολαία το erasmus την απασχόληση την έρευνα την καινοτομία και σας ρωτώ κύριε Κάνης, ως εκπρόσωπο του Συμβουλίου αλλά και ως παλιό Ευρωβουλευτή γιατί έχετε πετάξει στα σκουπίδια τις προτάσεις της Επιτροπής Μόντι για την αύξηση των ιδίων πόρων. Πώς μπορεί να προχωρήσει η πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης η οικονομική ολοκλήρωση της ονε η νομισματική ενοποίηση χωρίς να κοιτάμε το κοινωνικό θέμα. Κύριε Γιούνκερ και κύριε Κάρινς, στο Γκέτεμπορκ εγκρίθηκε η κοινωνική ατζέντα, αλλά παραμένει μια απλή ετικέτα. Δεν έχει αποκτήσει περιεχόμενο. Και όσο αυξάνονται οι ανισότητες, θα κερδίζει έδαφος ο λαϊκισμός των ακροδεξιών που θέλουν να διαλύσουν και την ευρώπη και τη δημοκρατία. πριν 80 χρόνια οι πολιτικοί πρόγονοι του κυρίου σαλβίνη της κυρίας λεπέν του κυρίου όρμπαν που κα, κακώς τον κρατάτε κύριε βέμπερ με αναστολή στις γραμμές του ευρωπαϊκού λαϊκού κόμματος οδήγησαν στο φασισμό και τον ναζισμό και σε έναν πολύ νεκρό πόλεμο. αν θέλουμε λοιπόν να υπερασπίσουμε τη δημοκρατία πρέπει στις επόμενες ευρωεκλογές να αποκτήσει μια ισχυρή πλειοψηφία μέσα στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο η άποψη που λέει ότι χρειαζόμαστε μια περισσότερο ενωμένη πολιτικά δημοκρατική και κοινωνική ευρώπη που να μειώνει τις ανισότητες και να μην τις αυξάνει. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λάμπερτς από την ομάδα των Πρασίνων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ. Καλώ ήλθατε πίσω στο Κοινοβούλιο, το οποίο το γνωρίζετε πολύ καλά. Πάντοτε δεν συμφωνούσαμε στι οικονομικέ υποθέσει, αλλά πάντοτε ήμουν πολύ εντυπωσιασμένο από τη δέσμευσή σα για το κοινοευρωπαϊκό πρόγραμμα. Και σήμερα είδαμε μια σχετική μαρτυρία. Και ε, πραγματικά ε, είναι τυπική δέσμευση αυτή που βρίσκουμε στι δημοκρατίε τη Βαλτική. Πιστεύω ότι οι χώρε του Μπενελούξ με τι τρει χώρε τη Βαλτική θα πρέπει να συνεργαστούν βαθύτερα. Γιατί αν μπορούν να βρουν συμφωνίε μεταξύ του, νομίζω ότι θα μπορούσαν να οικοδομήσουν γέφυρε και να προωθήσουν την ενότητα στην Ευρώπη, ίσω καλύτερα από το γαλλογερμανικό ντουέτο που φαίνεται αυτή τη στιγμή να είναι κάπω τσακωμένο. Μου άρεσε πάρα πολύ η ομιλία σα μου άρεσε που μας υπενθυμίσατε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ε, ένα project ειρήνης ε, και χρησιμοποιεί περισσότερο το διάλογο παρά τη βία. Αυτό είναι αιτιολόγηση όχι τον περασμένο αιώνα, αλλά η σημερινή αιτιολόγηση του ευρωπαϊκού οικοδομήματος ε, και μου άρεσε και η μεταφορά με το δεμάτι. Όπως και εσείς έρχομαι από μικρή χώρα, αλλά και μεγάλες χώρες και μου άρεσε αυτό που είπατε για την ενιαία αγορά. Η ενιαία αγορά είναι η έσχατη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, γιατί παρόλο ε, που έχουμε τέτοιες συμφωνίες διέπονται από τους δημοκρατικούς θεσμούς, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αλλού δεν ε, το βρίσκεται σε άλλε συμφωνίε ελευθερών συναλλαγών. Επίση, ε, μου άρεσε ε, το θέμα τη ήταν κάθετο για την νομοποίηση παράνομων εσόδων. Και μα αρέσει να ακούμε αυτό το λόγο, γιατί ξέρω ότι είστε ισχυρά δεσμευμένο για το θέμα αυτό. Επίση, θα ήθελα επίση να διαφωνήσω, όχι απαραίτητα με όσα είπατε, αλλά με κάποιε δράσει και θέσει τη κυβέρνηση τη Λετωνία. Καταρχήν, για μα του Πρασίνου, το Ευρωπαϊκό Κοδόμα θα πρέπει να αποτελέσει τη μηχανή, να έχει την ηγετική θέση τη οικονομική μετάβαση στις κοινωνίε μας. Αν δεν μπορέσουμε να τι κάνουμε να ταιριάξουν με τα όρια που μα θέτει η φύση, ε, απειλείται η ύπαρξη τη ίδια ανθρωπότητα. Είναι επίση θέμα ηγεσία. Αν εμεί η Ευρώπη δεν έχουμε ηγετική θέση σε αυτή τη μετάβαση, άλλοι θα το κάνουν. Και τότε εμεί ε, θα μείνουμε με το να αγοράζουμε τι δικέ του λύσει, παρά να δίνουμε τι δικέ μα στον υπόλοιπο κόσμο. Ε, μια περίπτωση και τον φέρετε, είναι η γεωργία. Η κοινή αγροτική πολιτική είναι ο μεγαλύτερο προπολογισμό τη Ένωση. Θα πρέπει κάθε λεπτό του ευρώ που δαπανάται σε αυτό αυτή να συνεισφέρει στην μεταμόρφωση του γεωργικού μας μοντέλου, έτσι ώστε να μειώνονται οι εκπομπές διοξείδου του άνθρακα, να αποκαθίσταται η ποιότητα του εδάφους και η βιοπικιλότητα. Η κοινή γεωργική πολιτική προωθεί ένα προτεκτηριστικό μοντέλο που καταφέρετε ε, κατά αυτόν τον στόχο και η κυβέρνησή σα ε, το υποστηρίξει και θεωρείτε ότι είναι πολύ πράσινο για τα γούστα σα. Καταλαβαίνω ότι η χώρα σα και συμφωνώ θέλει το δικό τη μερίδιο τη ε, ΚΑΠΟ Όμω είμαστε πεπισμένοι ότι ο καλύτερο τρόπο να επιτευχθεί αυτό ο στόχο είναι να αγωνιστείτε για μια πιο πράσινη κοινή γεωργική πολιτική που απομακρύνεται από αυτό το πρωτοκριστικό μοντέλο και τη βιομηχανική γεωργία. Η δεύτερη πτυχή έχει να κάνει με την ηθαγένεια. Αναφέρεται τι ευρωπαϊκέ αξίε και αν διαβάσετε το άρθρο 2, η πρώτη αξία που αναφέρεται εκεί είναι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια δεν ε, μπορεί να διαιρεθεί. Αφορά ε, όλους τους ανθρώπους και σήμερα και στο μέλλον. Η ε, Λετωνία, καθώς ανήκει χωρίς να θέλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει καταλήξει στο να είναι σημαντικό μέρος της Σοβιετικής Ένωσης. Έχει καταλήξει να έχει πάρα πολλούς Πολίτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση όμω ε, δεν πρέπει να διατηρεί απάτριδε 10% του πληθυσμού. επίση. Ε, πρέπει να ε, κάνετε περισσότερα, να προωθείτε τα δικαιώματα των μενοτήτων και να καταπολεμείτε τι διακρίσει κυρίω σε ό,τι αφορά τι αναπηρίες, την ηλικία ή το γενετήσιο προσανατολισμό. Τρίτον, καλώ ορίζουμε και σήμερα καταφέρετε να το αποφύγετε αυτό ότι και οι τρει δημοκρατίε τη Βαλτική έχουν αποφύγουν την ταξική στάση που έχουμε δει στο θέμα του ασύλου και τη μετανάστευση. Πραγματικά εκτίμησα τα λόγια για σας στο θέμα αυτό. Παρ' όλα αυτά, πρόσφατα η κυβέρνησή σα ε, δήλωσε ότι είναι αντίθετη σε οποιοδήποτε δεσμευτικό ε, σχέδιο μετεγκατάσταση, το οποίο μόνο αυτό θα οργανώσει την Ευρωπαϊκή Ελληνική. Επίση, αρνήθηκε να υπογράψει το Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΙΕ για τη μετανάστευση, το οποίο απλώ ε, παρέχει κατευθυντήριε γραμμέ για το πώ θα αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση. Και εγώ και εσεί γνωρίζουμε ότι δεν είναι νομικά δεσμευτικό και βασίζεται σε αξίες ε, για τον επιμερισμό της ευθύνης, ε, της μη εισαγωγής διακρίσεως και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αναγνωρίζει ότι μόνο μια συνεργατική προσέγγιση θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση. Θα πρέπει όμως η Λετωνία να υπογράψει το έγγραφο αυτό. Και καθώ πλησιάζουν οι ευρωεκλογέ, αυτή είναι η τελευταία συζήτηση για το μέλλον τη Ευρώπη σε αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βασιστείτε σε εμά για να υπερασπίσουμε ακούραστα την ε, πρώτη ε, προσπάθεια για να οικοδομήσουμε μία ε, διεθνική δημοκρατία. Επίση, βασιστείτε σε εμά για να την κάνουμε να λειτουργήσει για όλου, θέτοντα ε, στο επίκεντρο την οικονομική αξιοπρέπεια παρά τα οικονομικά κέρδη. Μία πιο ελεύθερη, βιώσιμη και δημοκρατική Ευρώπη είναι αυτό που θέλουν οι πολίτες ε, και εμείς θα ζητήσουμε τη δική τους εμπιστοσύνη ακριβώς για να παράξουμε αυτό το αποτέλεσμα. Και εξ ε, του EFDD, παρακαλώ κύριο Ευχαριστώ, αγαπητέ Πρόεδρε. Κύριε Πρωθυπουργέ Κάριντς, αξιότιμε αντιπαλέ μου, ο Ζαν-Κλοντ Γιούγκερ, πρώτα απ' όλα σας εύχομαι καλό Πάσχα για το Πάσχα που έρχεται και να σας πω και τα εξή. Όλο αυτό το επεισόδιο με την Παναγία των Παρισίων δείχνει τελικά πόσο λίγο μας ενδιαφέρει η πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης η ενότητα στην Ευρώπη που βασίζεται στην ελληνική φιλοσοφία, στο ρωμαϊκό δίκαιο, τη χριστιανική πίστη και την δημοκρατία θα έλεγα. Τελικά μας οδήγησε στη συνθήκη της Λισαβόνας και διαγράφηκε εκεί οποιαδήποτε μνήα στην χριστιανική Ευρώπη. Κάτι το οποίο όμως είναι ξένο προς την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με το σχέδιό της αυτό για ε, κοσμική Ευρώπη έχει απορρίψει ουσιαστικά την ίδια τη δικιά μας πολιτιστική κληρονομιά και μας οδήγησε έτσι σε πολιτιστική αδυναμία, κάτι το οποίο καταδικάζουν όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ευρωπαϊκό οικοδόμημα είναι ένα τρομακτικό οικοδόμημα καλτ ο Ροβεσπιέρος το είχε πει επίσης και με κάθε σεβασμό είπατε ότι η Ρωσία κάποια σχέση έχει με το Brexit. Μα συγγνώμη κύριε, οι Βρετανοί το 1940 πολέμησαν τον αυταρχισμό και είναι σε θέση να αποφασίζουν από μόνοι τους για το τι θέλουν ή δεν θέλουν από την Ευρώπη. Και δεν θέλουν γραφειοκρατικό αυταρχισμό από την Ευρωπαϊκή Γραφειοκρατία. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι αλήθεια ότι είναι ε, μοναδικό, γιατί θέλει να είναι κυρίαρχο και το δικό μας, στο δικό μας κοινοβούλιο κυριαρχεί μία ελίτ η οποία για πάνω από 30 χρόνια ηγείται από αυτούς τους Eurocult εύκολα μπορούμε να πούμε ότι φεύγουμε, ακολουθούμε τους κανόνες του ΠΕ και τίποτα άλλο. Αλλά οι Eurocalls αποφάσισαν διαφορετικά και αποφάσισαν, όπως η Πρωθυπουργό μας, να οδηγήσει την χώρα μας σε τόσες περιπέτειες. Ακούμε πολλές ανοησίες για διάφορα backstop στην Ιρλανδία και ότι τελικά μας απειλεί η Ευρώπη. Και αυτή η ευρωλατρεία μας έχει οδηγήσει εδώ που μας έχει οδηγήσει. Η κυρία Μέη αδίκως έχει αναγκαστεί να οδηγηθεί σε μια